Liebe Αγαπητοί συνάδελφοι, παραλαμβάνει τη συνεδρίαση και το πρώτο θέμα στην μέρη σε διάταξη είναι η έκθεση της κυρίας Κόμη κατά πολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. Και θα δώσω το λόγο πρώτα απ' όλα στην κυρία Κόμη 4 λεπτά. Πού είναι? Πού είναι? Μα Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, θα την ψάξουμε. Αλλά επειδή έχουμε πολύ φόρτο εργασία, θα πρότεινα, αν η κυρία Επίτροπο ε, Μπιενκόφσκα είναι διατεθειμένη, να ξεκινήσει εκείνη. Παρακαλώ, κυρία επίτροπο έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καθυστερήσεις πληρωμές λοιπόν. Ξέρουμε ότι είναι πολύ σημαντικό θέμα. Η καθυστέρηση στις πληρωμές δημιουργεί πρόβλημα που έχει τεράστια επίπτωση στις ε, επιχειρήσεις μας. Να επενθυμίσω το ιστορικό του θέματος. Ξεκινήσαμε το 1995 με συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ε, περιόδους πληρωμών, για τις εμπορικές συναλλαγές και είπαμε ότι οι καθυστερήσεις ήταν κίνδυνος για την επιβίωση των επιχειρήσεών μας. Το 2000 είχαμε την πρώτη οδηγία για τις ε, καθυστερημένες πληρωμές, αλλά η κατάσταση δεν βελτιώθηκε. Αντίθετα, οπότε το 2011 είχαμε μια αναθερωμένη οδηγία με πιο αυστηρούς κανόνες για να καταπολεμηθούν οι καθυστερήσεις και από δημόσιους και από ιδιωτικούς φορείς. Το 2016 η έκθεσή μας για την εφαρμογή της οδηγίας σημείωσε ότι μειώθηκε η μέση καθυστέρηση. Μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι ε, έχουμε ξεπεράσει το πρόβλημα. Βεβαίω όχι. Υπενθυμίζω, μόνο μία στις τέσσερις επιχειρήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο πληρώνει εντός ε, της ε, περίοδου συμβατικής υποχρέωσης. Δηλαδή 60% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων πληρώνονται τακτικά καθυστερημένα. Και αυτό είναι πραγματικά επικίνδυνο. Πάνω από τις μισές επιχειρήσεις υφίστανται καθυστερήσεις άνω των 90 ημερών για μια μικρή εταιρεία αυξάνεται η δυνατότητα πτώχευσης μετά από έξι ημέρες ε, καθυστέρησης. Και γι' αυτό οι καθυστερημένες πληρωμές είναι υπεύθυνε για 25% των ε, πτωχεύσεων στην Ένωση. Όπως παντού στην οικονομία, η καθυστέρηση πληρωμών ιδιαίτερα θίγει τι μικρομεσαίες που ε, χρειάζονται μόνιμα ρευστότητα για να μπορούν να λειτουργούν φταίει εν μέρη η πλήρωση οδηγία. Όχι, δεν νομίζω. Συμμερίζομαι την άποψη της εισηγήτριας ότι η οδηγία είναι το πιο κατάλληλο μέσο για να καταπολεμηθούν αυτές οι καθυστερήσεις. Η Επιτροπή μας εφήρμοσε αυστηρά την οδηγία. Από τη μία έχουμε ξεκινήσει ενεργό διάλογο με τα κράτη-μέλη, δώσαμε κατευθυντήρες γραμμές, ανταλλαγή ε, βελτίστων πρακτικών, αλλά από την άλλη μεριά δεν διστάσαμε να έχουμε και πιο αυστηρά και ε, επίσημα μέτρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν έξι περιπτώσεις διαδικασιών επί παραβάσεις στην Ένωση. Εν εξελίξη. Σύντομα θα πρέπει να δούμε την αναθεώρηση. Όχι, ε, είναι ακόμη νωρί για να δούμε ε, αν χρειάζεται περαιτέρω αναθεώρηση. Είναι περίπλοκο το θέμα, δεν αρκεί η νομοθεσία για να επιληθεί. Θεωρώ ότι οποιαδήποτε αλλαγή είτε του αυστηρού είτε του ήπιου νόμου πρέπει να ακολουθήσει μία αλλαγή στην οτροπία των, διοικη, των επιχειρήση. της επιχειρήσης. Πολλές φορές οι καθυστερήσεις αυτές είναι ηθελημένες. Ξέρουμε πολύ καλά ότι κάποιες επιχειρήσεις ε, δεν πληρώνουν τους προμηθευτές τους, γιατί αυτό είναι ένας δωρεάν ε, τρόπος ε, δανεισμού στην ουσία. Αλλά έχει κόστος, έχει κόστος για όλους μας, για την οικονομία. έχει κόστος στην πραγματική οικονομία. Διότι ε, οι καθυστερήσεις αυτές μετά έχουν ε, ένα, δημιουργούν ένα φαινόμενο ντόμινο. Ο προμηθευτής δεν πληρώνει τον περαιτέρω προμηθευτή και ούτω καθεξής. Μετά ξεκινάνε μακροσκελείς ε, διοικητικές υπηρεσίες που τεχνητά επιμηκύνουν την καθυστέρηση. Αυτό ιδιαίτερα όπως είπα και πάλι θίγει ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις ε, δημόσιες αρχές. Οι δημόσιες αρχές που καθυστερούν είναι ακόμη πιο ασυγχώρητες από ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Γιατί θα πρέπει να θυμηθούμε ότι αυτές οι ίδιες δημόσιες αρχές έχουν ελάχιστη ανοχή όταν τους οφείλονται από τις επιχειρήσεις ποσά. Για παράδειγμα, οι εφορίες. Πολύ επικίνδυνα όλα αυτά. Η έκθεση καταδεικνύει ότι πόσο φοβούνται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πολλές φορές φοβούνται οι επιχειρήσεις να εφαρμόσουν τα δικαιώματα που έχουν ε, μέσω της οδηγίας. Δέχονται αθέμητες ε, συνθήκες πληρωμής ε, από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Η κατάχρηση γίνεται συνήθεια, η συνήθεια γίνεται νοοτροπία. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει ελευθερία συμβατικής διαπραγμάτευσης αλλά αυτό δεν θα πρέπει να αξιοποιείται σε βάρος των ε, επιχειρήσεων ε, που τους οφείλονται ποσά. Πρέπει να υπάρχει σωστή ισορροπία μεταξύ της καταπολέμησης των καθυστερήσεων και της διατήρησης της συμβατικής ελευθερίας. Πρέπει επίσης να είναι πιο διαφανείς οι πρακτικές αυτές, να υπάρχουν ισχυρότερες ε, πολιτικές εφαρμογής του νόμου και αλλαγή της νοοτροπίας των μικρομεσαίων. Χαίρομαι που η έκθεση περιέχει διάφορα πορίσματα της έκθεσης εφαρμογή της δικής μας από το 2016. Μπορούμε να επιτύχουμε πολύ περισσότερο εάν ε, δίνουμε πάντα το παράδειγμα. Μπορούμε να είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί. Η οδηγία καλεί να αλλάξει εντελώς οτροπία μας όσον αφορά τις πληρωμέ. και κατά τη γνώμη μου αυτός πρέπει να είναι ο ίστατος στόχος μας. Οι ταχείες πληρωμές επιταχύνουν τη λειτουργία της οικονομίας και ωφελούν τους πάντες στην οικονομία. Συγχαίρω την έκθεση για το ισχυρό μήνυμα που στέλνει και για τις ε, αμοιβέ που δίνει προς τις ταχείες πληρωμές. Τέλος, η συγγήτρια, η κυρία Κόμη, εργάστηκε πολύ σκληρά, αλλά και η Ήταν, ήταν τεράστια προσπάθεια, σε σύντομο χρονικό διάστημα, το αποτέλεσμα είναι μεθοδικό, ισορροπημένο, εμπνευσμένη έκθεση. Ευχαριστώ και τον πρόεδρο Ταγιάννη, που ήταν ο προκάτοχός μου, γιατί εκείνος ενέκρινε και άρχισε να εφαρμόζει την οδηγία. Προσβλέπω στην περαιτέρω συζήτηση και σας καλώ να την εγκρίνετε αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια. Την κυρία Κόβλη. Πρόεδρε, καταρχά να ζητήσω συγγνώμη γιατί είχα καταλάβει ότι στις 6 θα ξεκινούσε η συζήτηση. Ζητώ συγγνώμη από τους συναδέλφους και ιδιαίτερως από την Επίτροπο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω κυρίως τους συναδέλφους που συνεργάστηκαν μαζί μου για την σύνταξη της έκθεσης αυτής. Ένα πολύ σημαντικό θέμα, ένα πολύ ευαίσθητο θέμα και χρήσιμο για την επιβίωση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Το πρώτο αίτημα το οποίο έχει τεθεί είναι το από τι εξαρτάται η υγεία μιας επιχείρησης. Ήταν υπάρχει μια ισορροπία βέβαια ανάμεσα στο οικονομικό κομμάτι, στο κομμάτι το ιδιοκτησιακό και στο κομμάτι το παραγωγικό και αν μπορεί πραγματικά η επιχείρηση να προσφέρει και στην οικονομία στην οποία κινείται εθνική και διεθνή. Πολύ συχνά όμως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι το βασικό δίκτυο της βιομηχανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουν, συγγνώμη, πάρα πολλά προβλήματα απέναντι στην κρίση λόγω των καθυστερήσεων από πλευράς άλλων επιχειρήσεων και κυρίως από πλευράς του δημοσίου. Έξι στις δέκα πληρωμές πληρώνονται με καθυστέρηση παραβιάζοντας τη συμφωνία το 62% των περιπτώσεων οφείλονται σε οικονομική δυσκολία αυτών οι οποίοι χρωστούν. Ένα άλλο ποσοστό είναι εσκεμμένες καθυστερήσεις, 40% είναι διοικητικές γραφειοκρατικές δυσκολίες και 19% είναι ε, αντι, αντιπαραθέσεις και εμπορικές διαφορές και αυτό ε, οδηγεί και στη δημιουργία κυρίαρχων θέσεων για κάποιες από τις επιχειρήσεις εις βάρος των άλλων. Αν μπορούσε να υπάρχει σωστός τρόπος πληρωμών, τότε θα μπορούσαμε να αποφύγουμε τέτοιου είδους φαινόμενα, γιατί είδαμε ότι πολλοί επιχειρηματίες φτάνουν μέχρι την αυτοκτονία στην Ιταλία και σε άλλες χώρες. Είναι τόσο, θα έλεγα, απελπισμένοι ε, και δυστυχώς ε, καταλήγουν ε, λόγω της μη πληρωμής ε, αυτών που τους οφείλουν. Ο στόχος τον οποίο είχαμε θέσει σε όλα τα κράτη-μέλη δεν έχει επιτευχθεί. Συνεπώς λοιπόν θεωρήσαμε να συμπεριλάβουμε στην πρόταση αυτή μια μεγαλύτερη προσπάθεια για να γίνεται η πληρωμή μέσα στον μήνα όπως είχε αποφασιστεί να υπάρχει μια μεγαλύτερη ασφάλεια σε σχέση με τη συμπεριφορά στις περιπτώσεις καθυστέρησης, να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες όπως και την δημόσια διοίκηση και να δημιουργήσουμε μια λευκή ε, βίβλο με αυτούς οι οποίοι είναι τακτικοί ε, πληρωτές έτσι ώστε να βοηθήσουμε γιατί πάρα πολλές μικρομεσαίες και startup ε, χάνουν ε, γενικά την ύπαρξή τους την ίδια λόγω των καθυστερήσεων και επίσης να προσπαθήσουμε να βρούμε και αντίμετρα σε επίπεδο φορολογικό, κάτι όμως το οποίο στη δική μου χώρα σαν παράδειγμα δεν γίνεται. Να προωθήσουμε τις ε, επιτυχημένες πρακτικές όπως την της Ισπανίας, που περιλαμβάνεται στην πρόταση όταν μια τοπική αρχή δεν είναι σε θέση να πληρώσει τότε παρεμβαίνει εκ μέρους της ε, η κρατική διοίκηση. Υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν λύσεις και στους δημόσιους διαγωνισμούς. Θα πρέπει να εξαιρούνται ε, κάποιοι εργολάβοι όταν δεν πληρώνονται από τον ή από πλευράς της συγκεκριμένη εταιρεία. Θα πρέπει λοιπόν να εφαρμοστεί η αρχή, όποιος κάνει λάθος πρέπει να το πληρώνει σε όλα τα επίπεδα. Και θα πρέπει επίσης να ανεβάσουμε το επίπεδο παρέμβασης των ενδιαμέσων διαιτητικών υπηρεσιών. Ε, γενικά πρέπει να το κάνουμε αυτό, μπορούμε να το κάνουμε και νομίζω ότι χάρη στην προσπάθεια όλων έχουμε μια καλή έκθεση. Ευχαριστώ κύριε Κυρία Κόμη, ο κύριος Πρέντα ε, έχει ζητήσει μια μπλε κάρτα, τη δέχεστε. Παρακαλώ κύριε Πρέντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να παρέμβω για να ρωτήσω γιατί η Ρουμανική Προεδρία δεν είναι παρούσα. Η κυρία Κόμη απευθύνθηκε στα κράτη-μέλη. Αλλά και κατά την προηγούμενη συζήτηση, τερικάμπρας, Μιλούσαμε για τα θεμελιώδη δικαιώματα και η Ρουμανική Προεδρία του Συμβουλίου απουσίαζε. Δεν κατάλαβαν ότι πρέπει να συμμετέχουν από πλευρά του Συμβουλίου σε αυτέ τι συζητήσει. Το θεωρώ απόλυτα λυπηρό. Θα ήθελα να καταλάβω τι γίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κόμη. θα αναζητήσω το λόγο, αλλά είναι πραγματικά αδικαιολόγητη η απουσία τους. Είναι μια έλλειψη σεβασμού απέναντι στους Ευρωπαίους πολίτες και τους Ευρωπαίους επιχειρηματίες. Ε, Διαπιστώνω ότι πολλές ε, προεδρίες ε, απουσιάζουν επανειλημμένα. Δεν είναι καλό. Αλλά επίσης δεν είναι καλό να κατηγορεί κανείς μόνο μία και όχι όλες τις προεδρίες. Νομίζω ότι οι συνάδελφοι θα πρέπει να αντιμετωπίζουν ισότιμα όλες τις προεδρίες. Τώρα έχουμε τους ομιλητές των πολιτικών ομάδων. Πρώτα απ' όλα για το ΕΛΚΟ κύριος Σφάμπ. μισή λεπτό. Ευχαριστώ. Συγχαίρω την εισηγήτρια. Κύριε Πρόεδρε, με ξέρετε. Ξέρετε ότι εγώ επανειλημμένα και σε άλλες προεδρίες έχω τονίσει την απουσία τους. Άρα δεν ισχύει αυτό που είπατε. Έχουμε μεγάλα προβλήματα στην Ευρώπη. Οι καθυστερήσεις μεταξύ Βορρά και Νότου είχαν μια διαφορά μεταξύ 100, που έφταναν ακόμη και τις 180 μέρες. Άρα υπάρχει περιφερειακό πρόβλημα. Γι' αυτό η έκθεση της κυρίας ε, Κόμη τα έλαβε υπόψη αυτά. Γιατί είδαμε την αλλαγή της οδηγίας για τις καθυστερήσεις που αποφασίσαμε στην προηγούμενη θητεία, όντως επιτύχαμε ορισμένα πράγματα. Η καθυστέρηση έχει μειωθεί. Αλλά οι καθυστερήσει αυτέ εξακολουθούν να αποτελούν πρόβλημα. Πρέπει να το δούμε γενικότερα στα πλαίσια τη ανάπτυξη τη οικονομία. Και αυτό το κάνει πολύ σαφέ η κυρία Κόμη. Οι μικρομεσαίε κυρίω ε, θίγονται. Και γι' αυτό απαιτεί η έκθεση ουσιώδη στοιχεία προς αυτή την κατεύθυνση. Και επίσης οι μικρομεσαίες θα πρέπει να ε, υπόκειται σε ορισμένες εξαιρέσει. Εάν κάποιες μικρομεσαίες ε, θέλουν να συμφωνήσουν κάποιες εξαιρέσει, θα πρέπει να επιτρέπεται, γιατί υπάρχει ελευθερία συμβατικής διαπραγματεύση και είναι διαφορετική η κατάσταση, αλλά ε, δεν σημαίνει αυτό ότι θα πρέπει να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των διαφόρων κλάδων τη οικονομία. Όπω και για τι αεροπορικέ εταιρείε, για όλε τι εταιρείε ισχύουν τα ίδια τα δικαιώματα των επιβατών, έτσι και εδώ πρέπει να ισχύουν οι ίδιε προθεσμίε. Ευχαριστώ για του σοσιαλιστέ. Η κυρία Γκραπίνη, 1,5 λεπτό. Ναι, κύρια Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας πω ότι ως η συγγήτρια του, του πολιτικής μου ομάδας Είχαμε μια ατμόσφαιρα πάρα πολύ ευχάριστη, δεν είχαμε καμία τριβή. Η κυρία Κόμη ε, προείδρευσε των συζητήσεων, τις ε, κατεύθυνε και η οδηγία που ήταν ένα πρώτο βήμα ε, δεν πέτυχε το στόχο, δηλαδή την μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών τη μεικτή ομάδα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπου είχαμε αυτή τη συζήτηση, ότι όλοι παρουσίασαν το ίδιο πρόβλημα, όλα τα κρατημέλη, ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν αρκετή διαπραγματευτική ισχύ ε, στις ε, διαπραγματεύσεις. Εκεί πρέπει να παρέμβουμε στις σχέσεις ε, με τις δημόσιες αρχές, το λέω και εγώ, θα πρέπει να υπάρχουν αποζημιώσεις. Δεν θα πρέπει η μικρομεσαία επιχείρηση να βρεθεί με ένα έλλειμμα λόγω των καθυστερήσεων. Ναι, Κυρία Επίτροπε, πρέπει να βελτιώσουμε την νοοτροπία της επιχείρησης, αλλά τι γίνεται με την νοοτροπία των δημοσίων αρχών που δεν πληρώνουν και καθυστερούν και αυτό είναι βλαβερό και για την ε, ταμιακή ροή των επιχειρήσεων. Ε, θα μπορούμε να διαπραγματευτούμε για μια λίστα λευκή ε, για να υπάρχει διαφάνεια, αλλά και μηχανισμός για να μπορούμε να αποφύγουμε τις πτωχεύσεις των μικρομεσαίων. Γι' αυτό πρέπει να τροποποιηθεί αυτή η οδηγία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γραπίνη. Ο κύριος Ζούμπιχ έχει μια μπλε κάρτα για σας. Συμφωνείτε, τη δέχεστε. Ναι, παρακαλώ, ο κύριος ε, Ρίμπη. Θέλω να ρωτήσω. Δεν θα ήταν δυνατόν να ασχοληθούμε και να δώσουμε διαφανή στοιχεία για τις καθυστερήσεις πληρωμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε πολλά προγράμματα όπου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις περιμένουν πολύ για να επανέλθει η ρευστότητά τους. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα κατάλογο στην Ένωση για να διαπιστώσουμε ότι και εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση τηρούμε την ε, ε, οδηγία αυτή. Ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα να πω ότι ο κύριος Ρούμπιτς είναι πάρα πολύ δραστήριος ε, στην ομάδα για τις μικρομεσαίες και για τα ενδιαφέροντά τους. Ναι, συμφωνώ, αυτό πρέπει να κάνουμε και ελπίζω, κύριε Επίτροπε, ότι αυτή η πρόταση του κύριου Ρούμπιτς θα ληφθεί υπόψη διότι υπάρχουν και ε, καθυστερήσεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη-μέλη καθυστερούν και αυτά με τη σειρά τους ε, να πληρώσουν τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ελπίζω αυτή η πρόταση να ληφθεί υπόψη. Ευχαριστώ πολύ. Για το ίσια ο κύριος και 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Η ελευθερία είναι βασική αρχή για τη σχέση μεταξύ επιχειρήσεων και διασφαλίζει φυσικά τη λειτουργία της οικονομίας. Οι δραστηριότητες ε, που θίγουν την διαπραγματευτική ελευθερία δεν επιτρέπονται. Γιατί αυτό σημαίνει ότι η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο παρεμβαίνουν στη σχέση μεταξύ ιδιωτικών ε, εταιριών. Γιατί οι πολιτικοί νομίζουν ε, ότι τα ξέρουν όλα. Πολύ καλύτερα από τις επιχειρήσεις. Και έχουν αυτή την τάση την έμφυτη να τα ρυθμίζουν όλα. Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μην παρεμβαίνουμε καθόλου. Φυσικά. Κάποιε εταιρείε καθυστερούν τι πληρωμέ του. Αλλά αφήστε την αγορά να το ρυθμίσει. Γιατί μετά δεν θα απευθυνθούν σε αυτού οι άλλε επιχειρήσει. Δεν μπορεί να τα κάνει η Κομισιόν αυτά. Δεν θα λειτουργήσει. Αν η Επίτροπο νομίζει ότι όντω πρέπει να ασχοληθεί η Επιτροπή, ε, ξεκινήστε τότε με τον εαυτό σας τον ίδιο. Γιατί πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημείωσε τεράστιες καθυστερήσεις με τις πληρωμέ τη. Όλοι οι ενωσιακοί πόροι εκταμιεύονται αργά και χωρί κανένα λόγο. Και το Κοινοβούλιο δεν λαμβάνει ε, εν ευθέτω χρόνο ε, τα ποσά που του οφείλονται. Μην ασχολείστε με τον ιδιωτικό τομέα. Κοιτάξτε τα του οίκου σα. Ευχαριστώ. Για την Άλντε, ο κύριος Ελίμοβιτς, δύο λεπτά. Ευχαριστώ. κυρία Πρόεδρε. Όλη η ευρωπαϊκή οικονομία κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις επηρεάζονται αρνητικά από τις καθυστερήσεις. Ε, έχετε βεβαίως υπάρχουμε και μερικές δράσεις, αλλά αυτό δεν αύξησε την ταμιακή ροή των επιχειρήσεων. Λίγο την αύξησε, έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε. Πάνω από τα μισά κράτη-μέλη Εκεί οι επιχειρήσεις ε, δεν ε, τηρούν τις 30 μέρες ε, που επιβάλλει ο νόμος και αυτές οι επιχειρήσεις, οι μικρές, δεν ζητούν αποζημιώσεις διότι φοβούνται να γίνουν ο εχθρός κάποιου που έχει τα χρήματα. Η έκθεση προτείνει μέτρα τα οποία θα βελτιώσουν την κατάσταση. Αν τα κράτη-μέλη να έχουν, να έχουν και αυτά αυστηρότερους ε, νόμους και χρειάζονται πληροφορίες ε, υποχρεωτικές ε, όπου λέχθηκε μια βάση δεδομένων μητρώα και για το δημόσιο και για τον ιδιωτικό τομέα κάνουμε έκκληση στα κράτη-μέλη να έχουν μια μεσολάβηση, ούτω ώστε αυτές οι επιχειρήσεις να μπορούν να απευθυνθούν σε κάποιον άλλον που να τις αντιπροσωπεύσει και να αγωνιστεί για αυτές. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να λάβουν όλα τα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι δημόσιες αρχές πληρώνουν εν ευθέτω χρόνο γέρος τους προμηθευτές. Καμιά φορά υπάρχουν οικονομικοί λόγοι, υπάρχουν όμως και πολιτικοί λόγοι. Κάνοντας το αυτό, τα κράτη-μέλη θα αυξήσουν ε, την, ε, τα, την ταμιακή ε, κατάσταση των επιχειρήσεων. Θα μπορούν και αυτές να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και το κλίμα των επιχειρήσεων θα βελτιωθεί πολύ περισσότερο από ό,τι είναι στη σημερινή κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τους πράσινους. Ο κύριος Σόλτες, δύο λεφτά. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα για την λειτουργία της οικονομίας στην Ένωση. Πρέπει να υπάρχει πειθαρχία με τις πληρωμές. Γιατί στο παρελθόν ε, καθημερινά διαπιστώναμε αυτές τις καθυστερήσεις. Και θίγουν πολλές επιχειρήσεις. Δεν είναι καλή κατάσταση στην Ένωση γιατί κυρίως οι μικρομεσαίες εφίστανται πίεση λόγω αυτής της καθυστέρησης. Γιατί κυρίως οι μικρομεσαίες ε, υφίστανται αυτού του είδους την ε, συμπεριφορά. Και πολλές ε, πτωχεύουν. Οπότε αυτό σημαίνει ότι οι οικογένειες των εργαζομένων τους θίγονται. Βεβαίως πολλά μπορεί να τα ρυθμίσει η αγορά. Αλλά χρειαζόμαστε και σαφείς κανόνες για να προστατεύσουμε τους αδύναμους από τους ισχυρούς και να αποφευχθούν οι καταχρήσεις από πλευρά των ισχυρών. Γιατί υπάρχουν αθέμητες εμπορικές πρακτικές, απαράδεκτες. Και η καθυστέρηση των πληρωμών είναι μόνο ένα στοιχείο αυτών των πρακτικών. Πολύ συχνά επιστρέφονται για παράδειγμα εμπορεύματα τα οποία δεν επολύθησαν από τον ε, περαιτέρω αγοραστή και οι μικροπρομηθευτές αντιμετωπίζονται σκιά. Πρέπει λοιπόν να έχουμε τους κατάλληλους μηχανισμούς για να αντιμετωπίσουμε και αυτά τα θέματα. Οι συνάδελφοι αναφέρθηκαν ήδη στις υπηρεσίες ε, διαμεσολάβησης, διαιτησίας. Αλλά, να πω και κάτι ακόμη. Ο δημόσιο τομέα επίση καθυστερεί τι πληρωμέ. Πολλά πρέπει να κάνουμε για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και των καθυστερήσεων των δημοσίων φορέων. Είναι ντροπή αυτά τα πράγματα. Οι δημόσιες αρχές να συμβάλλουν σε αυτές τις καθυστερείς πληρωμών. Ο κύριος Μαστάλκα για την ΚΟΕ. Ευχαριστώ πολύ. Κάθε χρονιά στην Ένωση χιλιάδες μικρομεσαίες πτωχεύουν. Λόγω των καθυστερήσεων πληρωμών Λόγω λοιπόν αυτής της καθυστέρησης έχουμε πτώχευση, κοινωνικά προβλήματα, ανεργία. Η οδηγία του 2011 στόχευε να βοηθήσει τις επιχειρήσεις. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για την αναλυτική περιγραφή που κάνει της κατάστασης. Για την εφαρμογή δηλαδή αυτής της ε, οδηγίας. Προέκυψε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά προβλήματα. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει επαρκής γνώση της δυνατότητας χρήσης αυτής της οδηγίας, δηλαδή άγνοια της οδηγίας. Μόνο ένα μικρό ποσοστό επιχειρήσεων είπαν ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση σε σχέση με την καθυστέρηση πληρωμών εναντί του. Πολλά μπορούμε να βελτιώσουμε. Συμφωνώ, μάλλον δεν συμφωνώ με τον συνάδελφο Ζιούλικ, δεν είναι σωστό να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά. Θα ήταν η χειρότερη αντιμετώπιση των μικρομεσαίων. Και κυρίως ε, αυτό που είναι ιδιαίτερα λυπηρό είναι οι δημόσιες αρχές να μην τι πληρώνουν. Έχει πλήρω τη στήριξή μου η συγγήτρια. Συμφωνώ με τι προτάσεις που κάνει για να εφαρμοστεί καλύτερα η οδηγία. Στόχο μα πρέπει να είναι δίκαιο ανταγωνισμός. Ισότιμες συνθήκε ανταγωνισμού για όλε τις επιχειρήσεις. Ίσως είναι η τελευταία φορά που παίρνω το λόγο εδώ στο Κοινοβούλιο. Οπότε ευχαριστώ όλους ε, ε, εκείνους με τους οποίους συνεργάστηκα και ευχαριστώ και τους υπαλλήλους και τους διερμηνείς. Ευχαριστώ πολύ. Σας εύχομαι, λέει Πρόεδρος, ε, πολλή, κάθε επιτυχία και τύχη στην περαιτέρω σταδιοδρομία σας. Λοιπόν, τώρα περνάμε στου επόμενους ομιλητές, η κυρία, Τουν, η Φόντουν Ουνχόλστάιν. Πρόεδρε, πάντα υποστήριζα ότι γενικά τα πράγματα βελτιώθηκαν στη χώρα μου από τότε ε, που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα μου. Αλλά δυστυχώς πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα. Αρκετά πετύχαμε βέβαια, όπως τον γεωγραφικό αποκλεισμό, το roaming, την περιαγωγή. Ε, και άλλα θετικά από τα οποία ωφελούνται οι Ευρωπαίοι πολίτες. Αλλά σήμερα συζητάμε την κατάσταση των επιχειρηματιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκεί τα πράγματα δεν είναι καλά. Πάρα πολλέ μικρομεσαίες λοιπόν αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω απλήρωτων ε, χρεών. Απειλούνται και από πτώχευση πολλές επιχειρήσεις γιατί οι επιχειρηματίες έτσι κι αλλιώς έχουν προβλήματα ρευστότητας, έτσι και αλλιώς έχουν προβλήματα φορολογικού τύπου και γι' αυτό βλέπουμε ότι η νομοθεσία από την οποία έχουμε περάσει δεν λειτουργεί με σωστό τρόπο. Η έκθεση λέγει ότι η νομοθεσία δεν εφαρμόζεται με τον σωστό τρόπο σε ορισμένες χώρες μέλη και αυτό είναι κάτι το οποίο ε, θα έλεγα δημιουργεί προβλήματα. Απαιτείται λοιπόν να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια σε σχέση με τις συμπεριφορές των τομέα των πληρωμών. Έτσι αυτοί οι οποίοι χρωστούν θα πρέπει να πληρώνουν πολύ γρηγορότερα. Όταν περάσουμε λοιπόν την καινούργια οδηγία θα πρέπει να το κάνουμε ισορροπώντας τα διαφορετικά συμφέροντα. Η αρχική στόχη της οδηγίας αυτής είναι η αύξηση των θέσεων απασχόλησης και η προστασία αυτών οι οποίοι είναι χρεωμένοι. Κλείνοντα, θα ήθελα να πω ότι οι, μικιο, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι σημαντικές για την οικονομία και πρέπει να τις φροντίσουμε. Μέχρι στιγμή έχουν τηρήσει το χρόνο τους ε, οι ομιλητέ και ομιλήτρες. Ε, παρακαλώ να συνεχίσετε έτσι γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα στη μέση διάταξη σήμερα. Ντάντι, 1,5 λεπτό. Πρόεδρε, Επίτροπε, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η οδηγία του 2011 λειτουργήσε σχετικά θετικά, τουλάχιστον μείωσε λίγο τον χρόνο αναμονής πληρωμής για τις επιχειρήσεις. Γνωρίζουμε όμως ότι το 95% των μικρομεσαίων δεν παίρνουν τα χρήματά τους στους προκαθορισμένους χρόνους και μερικές φορές η καθυστέρηση αυτή οδηγεί σε πτωχεύσεις. Νομίζω λοιπόν ότι η έκθεση αυτή την οποία θα εγκρίνουμε αύριο πρέπει να προτείνει ακόμα περισσότερα σημεία βελτίωσης για να αντιμετωπιστεί η μάστιγα αυτή. Πρώτον, θα πρέπει για τις επιχειρήσεις οι οποίες ε, έχουν χρήματα να παίρνουν από το δημόσιο να ανταλαμβάνουν τα χρήματα αυτά με μεγαλύτερη ταχύτητα. Δεύτερον, να υπάρξουν δωρεάν διαιτητικές υπηρεσίες οι οποίες να βοηθήσουν τις ε, μικρομεσές και να έχουν τα οικονομικά μέσα για να, που δεν έχουν τα οικονομικά μέσα για να αντιμετωπίσουν ε, ε ιδιαίτερα ακριβές δικαστικές ε, υπηρεσίες. Και τρίτον θα πρέπει να υπάρξουν φορολογικές ε, διευκολύνσεις για αυτούς οι οποίοι πληρώνουν έγκαιρα. Νομίζω ότι βλέποντας τα αποτελέσματα, τα όχι ιδιαίτερα λαβρά των τελευταίων χρόνων, ε, οι δυσκολίες είναι πάρα πολύ ψηλές. Θα πρέπει λοιπόν το σύστημα το επιχειρηματικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βοηθηθεί. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον εγγυήσεων, σταθερότητας έτσι ώστε να μπορέσουν να διεξάγουν τις δραστηριότητές τους με σωστό τρόπο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι αληθές ότι ε, οι καθυστερήσεις πληρωμών βλάπτουν πολύ τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, για να μπορέσουν να καινοτομήσουν, να προσλάβουν, ε, χρειάζονται ταμιακά χρήματα. Διότι όταν κανείς καθυστερεί τις πληρωμές, τους αφαιρεί το οξυγόνο τους η Επιτροπή θα πρέπει να υποστηρίξει τις μικρομεσαίες που είναι ε, η σπονδυλική στήλη της οικονομίας μας, να αφήσουμε ε, και να στην νομοθεσία μας αυτό πρέπει να απαγορεύεται. Δύο στις τρεις επιχειρήσεις δέχονται καθυστερήσεις πληρωμών, ενώ δεν θα έπρεπε να το κάνουν. Γι' αυτό το 2017 το δικό μου κόμμα κατέθεσε ένα σχέδιο νόμου για να υπάρχει μία μέγιστη προθεσμία για τις πληρωμές. Θα πρέπει η Ευρώπη ε, να στείλει ένα μήνυμα ισχυρό για να αποτρέψει αυτές τις καθυστερήσεις. Έχουμε κάτι στο τώρα. τέσσερι τέσσερις συνάδελφοι χωρίς το λόγο. Θα τους δεχτώ και τους τέσσερις. Πρώτος, ο κύριος Σέντρο Γεύσκη. Ένα λεπτό. Πράγματι το θέμα αυτό έχει μεγάλη σημασία και έχει μεγάλη σημασία γιατί θέλει να αντιμετωπίσει μια καταστροφή της καθυστερημένες πληρωμές είναι ο πιο φθηνός τρόπος να δανείζεται κανείς χρήματα αυτός ο οποίος καθυστερεί την επιστροφή και είναι κάτι το οποίο φυσικά κοστίζει πάρα πολύ ε, για αυτούς οι οποίοι περιμένουν την πληρωμή. Νομίζω ότι με τις προτάσεις αυτές εν πολλής μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι. Όταν εμείς ξεκινήσαμε την διαδικασία αυτή, μιλήσαμε για τις δικές μας καθυστερήσεις σε προγράμματα όπως το Εράσμους κτλ. Τέσσερα χρόνια μετά μπορούμε να πούμε ότι τουλάχιστον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια των πληρωμών της έχει βελτιώσει την αποδελεσματικότητά της και μπορούμε λοιπόν να κατηγορήσουμε άλλους τομείς και επιχειρήσεις που καθυστερούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χόουαρθ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τον εισηγητή και την Επιτροπή. Όσοι από εμά είναι ιδιοκτήτες μικρομεσαίους, ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις γνωρίζουν ότι τα προβλήματα για την κερδοφορία είναι η έλλειψη ρευστότητας και οι καθυστερήσεις. Πέρυσι οργάνωσα μία συνάντηση με την Ομοσπονδία Μικρομεσαίων του Ηνωμένου Βασιλείου για να βελτιωθεί η εφαρμογή της οδηγίας στο Ηνωμένο Βασίλειο για τις καθυστερημένες πληρωμές. Ταυτόχρονα ε, σε σχέση ε, με τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς το να συνδεθεί ε, το θέμα αυτό είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό και ταυτόχρονα θα πρέπει το δημόσιο να είναι υπόδειγμα και να πληρώνει εγκαίρως Επίση υπάρχει το θέμα των υποχρεωτικών προθεσμιών πληρωμών από πλευρά των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Όλα αυτά είναι επιμέρους θετικά βήματα. Θα πρέπει να ξεκινήσει τώρα μια νέα διαβούλευση δημόσια για ένα ακόμα γύρο ενίσχυσης της εφαρμογής της οδηγίας για καθυστερημένες πληρωμές. Κυρία Κινίτσι. Ευχαριστώ Πρόεδρε παρά την οδηγία του 2011 για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα οι μικρομεσές, αντιμετωπίζουν πάντα καθυστερήσεις ε, και όχι μόνο από πλευράς ε, της δημόσιας διοίκησης. Στην Ιταλία και όχι μόνο σε αυτήν βέβαια, το οικονομικό δίκτυο, αν θέλετε, αποτελείται κυρίως από μικρομεσές. Υπάρχουν ε, καθυστερήσεις στις πληρωμές, από τις μεγάλες επιχειρήσεις προς τις μικρές και δεν διαμαρτύρονται για να μην διαρρήξουν τις εμπορικές αυτές σχέσεις. Αυτό είναι αθέμητες δράσεις από πλευράς των μεγάλων επιχειρήσεων και δημιουργεί προβλήματα στις μικρομεσαίες, ιδιαίτερα στον τομέα των τροφίμων και των γεωργικών προϊόντων, φύγονται οι μικροί παραγωγείς, ιδιαίτερα σε έναν τομέα ο οποίος έχει τόσο υψηλές ανισότητες. Πρέπει να ξεκινήσουν λοιπόν εκστρατείε ευαισθητοποίηση σε σχέση με το χρόνο καθυστέρηση και με τα νομικά μέσα εναντίον των καθυστερήσεων. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να ισχύει και για τη δημόσια διοίκηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τελευταίος, ο κ. Μαριάς. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Οι καθυστερήσει στι εμπορικέ συναλλαγέ η μη πληρωμή δηλαδή έγκαιρα από πλευράς ιδιωτικών επιχειρήσεων δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στον ίδιο τον ιδιωτικό τομέα και φυσικά είναι μια διαδικασία που μπορεί να οδηγήσει σε πτωχεύσεις. το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως είναι να χρωστάει το δημόσιο διότι το δημόσιο είναι αυτό το οποίο απαιτεί από τους φορολογούμενους να πληρώσουν και όταν δεν πληρώνουν ή έχουν δυσκολία να πληρώσουν φόρους όπως είναι οι φτωχοποιημένοι από τα μνημόνια έλληνες τότε το κράτος κάνει κατασχέσεις κάνει κατασχέσεις στους λογαριασμούς κάνει κατασχέσεις στην περιουσία τους. όμως αυτό το κράτος το ελληνικό δημόσιο οφείλει αυτή τη στιγμή με στοιχεία του δεκεμβρίου του 2018, χιλιάδες ένα δισεκατομμύριο ευρώ στον ιδιωτικό τομέα. και ξέρετε γιατί τα οφείλει; διότι κρατάει τα χρήματα προκειμένου να πληρώσει τους δανειστές για να δημιουργήσει το περίφημο πρωτογενέ πλεόνασμα και αυτό το γνωρίζει η κομισιόν αλλά προτιμάει να πληρώνονται οι δανειστέ από το ελληνικό δημόσιο παρά να πληρώνει το ελληνικό δημόσιο τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Επίτροπο για να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλα τα μέλη για αυτή τη συζήτηση, αλλά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κυρίως διότι ε, θεωρείται το θέμα των καθυστερημένων ε, πληρωμών σημαντικό και ίσως η ψηφοφορία αύριο θα είναι κάτι το καλό για το θέμα αυτό. Σε σχέση με το θέμα αυτό, από το 1995 στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ακόμα πολλή εργασία που πρέπει να γίνει κυρίως στον τομέα των αλλαγών νοοτροπίας που λέχθηκε. Είναι κάτι που κάθε επιχείρηση, κάθε δημόσια αρχή πρέπει να κατανοήσει ότι είναι προς όφελός της ε, αυτές οι έγκαιρες, οι εμπρόθεσμες πληρωμές είναι προς όφελός τους. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι βεβαίως τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρώπη και οι επιχειρήσεις και οι δημόσιες αρχές στην Ευρώπη έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις βάσει αυτής της οδηγίας. Θα ήθελα λοιπόν να σας επισημάνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισήγαγε έναν κανόνα μηδενικής ανοχής ε, για τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι είναι κάτι το καινούριο και ότι θα οδηγήσει σε καλά αποτελέσματα στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ και βεβαίως για όλη την εργασία που έγινε ε, για τις ε, καθυστερήσεις ε, πληρωμών που θα είναι χρήσιμη. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά η κυρία Κόμη. Ευχαριστώ την Επίτροπο, ευχαριστώ και όσους πήραν το λόγο. Ήταν επικοδομητικός ο διάλογος, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες και τους πολίτες. Δύο σύντομες σκέψεις. Πρώτον, τη στιγμή κατά την οποία ένα κράτος δεν εφαρμόζει σωστά την οδηγία, τότε ξεκινάει, θα πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία επί παραβάση. Αυτό οδηγεί σε κυρώσεις οικονομικές και αυτό βλάπτει εκ νέου τους πολίτες. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, δηλαδή από τη μία το κράτος δεν πληρώνει και από την άλλη ο πολίτης πληρώνει ουσιαστικά αυτά τα οποία οφείλει να πληρώσει σαν πρόστιμο το κράτος όπως είπατε πριν από εσά, ο προκάτοχός σας ήταν ο πρόεδρος Ταγιάννη και πράγματι ε, έθεσε το θέμα του επίπεδου του 3% έτσι ώστε να αναγκάζεται να πληρώσει η δημόσια διοίκηση. Αυτός δεν είναι κανόνας βέβαια στην υπόλοιπη Ευρώπη και γι' αυτό η Ιταλία δεν έχει καμία δικαιολογία όταν το δημόσιο, το κράτος δεν πληρώνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και θα περάσουμε στη ψηφοφορία αύριο. Ευχαριστώ κυρία Συγήτρια. Ολοκληρώνεται η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο, όπως είπατε και εσείς μόλις τώρα. Και τώρα, το επόμενο θέμα. Έκθεση της κυρίας Κάπελ. Ετήσι έκθεση για την χρηματοοικονομική δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Και καλωσορίζω και τον Βέρναρ Χόια που είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Παρακαλώ καθίστε. Και να δώσω το λόγο καταρχάς το λόγο στην εισηγήτρια, την κυρία Κάπελ. Τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε Κατάινεν, ε, Πρόεδρε Χόια, σήμερα θα συζητήσουμε την ε, ετήσια έκθεση δραστηριότητας ε, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους Κιώδης, τους συντάκτες νομοδοτήσεων, τις επιτροπές που είχαν στην αρμοδιότητα, την ομάδα μου, τις ομάδες τους. Ευχαριστώ πολύ. Μέσα σε λίγους μήνες και με πραγματιστικό τρόπο έχουμε μια συνολική έκθεση για τη δραστηριότητα της τράπεζας το 2016 για την περίοδο 16-19 η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, βασίζεται στις αρχές της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ανάπτυξη στην ενέργεια, την υγεία, την κινητικότητα, τις ε, υποδομές της υπαίθρου, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις μέσα κεφαλαιοποίησης και την καινοτομία. Σε αυτό το χρονικό πλαίσιο Είχαμε και την 60η ε, επέτειο της ε, ΕΤΕ και σας ευχαριστώ πολύ για δραστηριότητά σας. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι ο μεγαλύτερος ε, πολυμερής δανειστής στον κόσμο. Σε 60 χρόνια δόθηκαν 1,13 εκατομμύρια σε πάνω από 160 χώρες. Πρέπει να είμαστε περήφανοι για αυτόν τον απολογισμό. Τα δάνεια αυτά έχουν την υψηλότερη αξιολόγηση ποιότητας. Έχει τριπλό α και ίδια τράπεζα και λόγω της συντηρητικής ε, διαχείρισης των κινδύνων ε, ε, επειδή τα, δηλαδή τα προβληματικά δάνεια είναι μόνο 0,3% είναι πολύ καλή λειτουργία. Έχει ένα πολύ καλό χαρτοφυλάκιο επενδύσεων. Αυτές είναι οι βασικές αρχές λειτουργίας της ΕΤΕΠ. Οι βέλτιστες πρακτικές λοιπόν. Και ναι μεν Είπαμε ότι οι χρηματοδοτήσεις έχουν πάει σε 160 χώρες, αλλά 90% έχουν πάει στις χώρες της Ένωσης. Δώσαμε 78 δισεκατομμύρια για την ε, καινοτομία και το περιβάλλον και τις μικρομεσαίες. Το τελευταίο χρόνο δώσαμε πάνω από 200 δισεκατομμύρια για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των περιφερειών. Πάνω από 700.000 μικρομεσαίες ε, πήραν χρηματοδότηση. Να κάνω μια παρατήρηση ωστόσο. Το 2017 το 1 τρίτο περίπου των ε, δάνειων δόθηκαν σε δολάρια. Χθε ε, είχαμε στο σώμα μα τα 20 χρόνια του ευρώ, την επέτειο, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νόμισμα στον κόσμο. Ίσως στο μέλλον, κύριε Πρόεδρε, να μπορούσατε να κάνετε περισσότερες επενδύσεις σε ευρώ και σταδιακά να μειώσετε τις, ε, επενδύσει και τι καλύτερα σε δολάρια. Το 2017 δώσατε 13,9 δισεκατομμύρια για την ε, ψηφιακή οικονομία και για να ε, κατασταθούν 36 εκατομμύρια εφιών ε, μετρητών. Πολλά δώσατε επίσης για τις ανανεώσιμες ενέργειες, για την ενεργειακή απόδοση, για τη βιολογική πολυμορφία, το καθαρό νερό, το καθαρό ατμοσφαιρικό αέρα, την βιώσιμη, τις βιώσιμες μεταφορές κτλ είστε ο μεγαλύτερος δανειστής πρασίνων δανείων και έχετε χρηματοδοτήσει πάρα πολλά ε, προγράμματα για την ε, καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Παίζετε λοιπόν μεγάλο ρόλο για την ε, εφαρμογή των στόχων του Παρισίου. Χρηματοδοτήσατε επιχειρήσεις με 29,6 δισεκατομμύρια. Εκατοντάδες μικρομεσαίων επιχειρήσεων με εκατομμύρια εργαζόμενους. Οι μικρομεσαίες και τα startup παίζουν μεγάλο ρόλο για την ευρωπαϊκή οικονομία. Οπότε η στρατηγική σας γι' αυτό και η συνεργασία σας για να αντιμετωπιστεί το χάσμα χρηματοδοτήσεων πολύ σημαντική. Επίσης, κάνατε μεγάλη προσπάθεια και μέσω του ΕΦΣΥ για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη επενδύσεων λόγω της κρίσης. Δόθηκαν πολλά ποσά και Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μόλτεραν και οπωσδήποτε θα είστε υπεύθυνοι και για το νέο πρόγραμμα InvestEU την επόμενη περίοδο. Ευχαριστώ κυρία εισηγητρία. Και τώρα από πλευράς ε, προϋπολογισμών Γαρδιαθάβαλε Ρουβιάλ. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Χόιερ. Εξ ονόματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών θα ήθελα να παρουσιάσω τα θέματα τα οποία πρέπει να περιλαμβάνονται στην γνωμοδότηση σχετικά με τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Λόγω έλλειψης χρόνου θα συγκεντρωθώ στα πιο σημαντικά. Το θέμα είναι να μπορέσει να ενισχύσει την επενδυτική της δραστηριότητα και στον δημόσιο τομέα και στον ιδιωτικό τομέα και έτσι να μπορέσει να λειτουργήσει αντικυκλικά λόγω, η οικονομία λόγω των επενδύσεων αυτών, κάτι το οποίο θα οδηγήσει και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας, με μακράς διάρκειας επενδύσεις. Είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό να ενισχυθεί η στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, να βελτιωθεί η ενημέρωση και η πρόσβαση στα προγράμματα της ε, Τράπεζας Επενδύσεων έτσι ώστε να μπορούν να συμμετέχουν με καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και όχι μόνο λόγω της ύπαρξης του ΕΦΣΥ ότι η συνεργασία με τις αναπτυξιακές εθνικές τράπεζες θα πρέπει να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο και έτσι θα αποκτήσουν μεγαλύτερη σημασία οι επενδύσεις και θα υπάρξει και μεγαλύτερη τεχνική βοήθεια. Και σχετικά τώρα με τις επενδύσεις προς ε, χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται μεγαλύτερη συνεργασία με τις αναπτυξιακές τράπεζες έτσι ώστε να είναι πιο αποτελεσματικές και να απομακρύνουν τις επικαλύψεις. Έτσι θα μπορέσουμε να πετύχουμε το 25% και ε, των επενδυτικών δυνατοτήτων σχετικά με την μετρίαση των συνεπειών των κλιματολογικών αλλαγών. Και θα ήθελα να ζητήσω επίσης ότι θα πρέπει να συνεχίσετε να εργάζεστε και να ε, επενδύετε έτσι ώστε να βελτιωθεί η διαφάνεια, ε, να υπάρχουν υπόλογοι και να ελέγχονται φυσικά και οι ενδιάμεσοι πληρωτές έτσι ώστε να αποτρέπονται περιπτώσεις απάτης. Με χαρά να δώσω το λόγο στον πρόεδρο της ΕΤΕΠ. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτέ, κυρίε και κύριοι, επιτρέψτε μου καταρχά να ευχαριστήσω την εισηγήτρια θερμότατα και του συνεργάτε τη για αυτήν την θαυμάσια έκθεση. Είναι μεγάλη χαρά που είμαι εδώ με εσά. Αυτή η συζήτηση παίζει σημαντικό ρόλο για την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και την ΕΤΕΠ. Πάρα πολλά θέματα που αναφέρονται στην έκθεση είναι πάρα πολύ χρήσιμα, ε, συναφή και εκτιμώ ε, τα όσα είπατε για το ρόλο της τράπεζας που είναι καταλήτης ε, για τις επενδύσεις και υποστηρίζει τις επενδύσεις, ε, την ανάπτυξη εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως επισημάνατε, ορθώς η ΕΤΕΠ είναι πάρα πολύ καλή και χρήσιμη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βάζουμε το χρήμα να δουλεύει όχι τόσο τα χρήματα των φορολογουμένων, αλλά τα χρήματα τα οποία συλλέγουμε από επενδυτές στην κέφαλη αγορά τα επενδυτικά σχέδια μας είναι μοναδικά. Τα κράτη-μέλη οφείλουν στην ΕΤΕΠ, αλλά δεν είναι η βασική πηγή χρηματοδότησης. Τα κράτη-μέλη εδώ και 60 χρόνια ε, πλήρωσαν μόνο 40 δισεκατομμύρια άμεσα σε χρήμα για να εξασφαλίσουν ε, το μερίδιό τους ε, στην κεφάλαιο της τράπεζας, τέσσερα καθενός. Και έτσι μπορέσαμε να εκματεύσουμε πάνω από 1,1 τρισεκατομμύρια όπως λέχθηκε ε, και έτσι έχουμε πάνω από 3 εκατομμύρια συνολικές επενδύσεις. Βλέπουμε την καλή αποτελεσματική χρήση των ευρωπαϊκών χρημάτων ακολουθούμε αυτήν την πολιτική. Χάρη σε εσά μπορούμε να, έχουμε, να εργαζόμαστε με τρόπο βιώσιμο ε, και ε, διαφανή. Έχουμε επίσης ε, και για το κλίμα, έχουμε πράσινα ομόλογα. Βιωσιμότητα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα όταν όλοι εγκομιάζουμε τα Ηνωμένα Έθνη που προσδιορίζουν τι είναι οι στόχοι της αηφόρου της διαρκούς ανάπτυξης βλέπουμε ότι ποτέ τα χρήματα των φορολογουμένων δεν θα μπορούσαν να μας επιτρέψουν να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους. Πρέπει να αντλήσουμε από τον ιδιωτικό τομέα, γι' αυτό ε, έχουμε αναπτύξει τα πράσινα ομόλογα και τώρα αναπτύσσουμε διάφορα ομόλογα τα οποία είναι ε, ευαίσθητα στην βιωσιμότητα. Επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ανακάμψει, αλλά η ανάκαμψη ε, είναι άνηση ανάμεσα στους τομείς και στις χώρες. Δεν πρέπει να είμαστε ποιικείς όταν ε, σκεπτόμαστε τα χάσματα, τα επενδυτικά, να σκεφτούμε τις ε, υποδομές. Βλέπουμε ότι έχει καθυστέρηση η Ευρώπη. Έχουμε το, το, το, το, εύση και σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια στο θέμα αυτό. Επίσης, έχει αναφερθεί η επιτυχία ε, του ΕΦΣΥ και ήταν ε, απόφαση του Κοινοβουλίου το πρόγραμμα αυτό να συνεχιστεί μέχρι το 2020 και και ήταν καλή απόφαση του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου να θυσιάσει 60 δισεκατομμύρια του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μεταφέρει από επιχειρήσεις στα σχέδια εγγύησεων και αυτή η άσκηση δεν είναι ίσως πάρα πολύ δημοφιλή ε, πράξη για έναν ε, βουλευτή, αλλά ήταν πάρα πολύ χρήσιμη από το Δεκέμβριο 2018 Έχουμε πάνω από 850.000 μικρομεσαίες που υποστηρίχθηκαν και ελπίζουμε 371,1 δισεκατομμύρια πρόσθετες επενδύσεις ε, θα προκληθούν. Βλέπουμε λοιπόν πώς μπορούμε να κάνουμε για να υποστηρίξουμε ε, τις, ε, τους σπάνιους δημόσιους πόρους και αυτή η μεταφορά που έγινε είναι καλό στοιχείο της πολιτικής σας θα πρέπει να κρατήσουμε από, την, το ΕΦΣΙ τα καλά στοιχεία για την εκπόνηση των μελλοντικών σχεδίων